να κάνουμε, να πετύχουμε αυτή την ισορροπία για να δοθεί το σωστό μήνυμα και στον υπόλοιπο κόσμο. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε κυρία Πίτροπε, Κλείνει εδώ, ολοκληρώνω τη συζήτηση για αυτό το σημείο. Θα ψηφίσουμε αύριο το μεσημέρι, 12.00 ώρα, την αντίστοιχη πρόταση ψηφίσματος που μας ε, υποβάλλει ο εισηγητής κύριος Παπαστάμκος. Και έτσι Περνάμε στο ακόλουθο σημείο στην ημερήσια διάταξη, που είναι και το τελευταίο αυτή τη ε, εκτενούς νυχτερινή συνεδρίασης ε, και είναι το σημείο το οποίο θα συζητήσουμε τώρα. Είναι η έκθεση του κυρίου Χόισλεϊν, το πρωτεϊνικό έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναζήτηση λύσεων για ένα παλαιό πρόβλημα. Έχει τον λόγο ο εισηγητής, ε, κύριος Χόισλεϊν, για τέσσερα λεπτά για να μας παρουσιάσει την έκθεσή του. Παρακαλώ κύριε Χόισλεϊν. Μάλιστα, Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχήν ευχαριστώ του κοιόδης εισηγητέ θερμά ε, για την αλληλέγγυα συνεργασία, συναδελφική συνεργασία για την έκθεση. Είναι μια φιλόδοξη έκθεση με τη μορφή που πήρε και θα ήθελα σύντομα να αναφερθώ στα σημεία που είναι σημαντικά. Και θα αναφέρω επίσης εξίσου και τα επίμαχα σημεία. Έχουμε τεράστιο έλλειμμα πρωτεϊνικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 80% της ανάγκης μας ε, το καλύπτουμε με εισαγωγές. Και η τάση είναι αυξητική δυστυχώς. Αυτό ανταποκρίνεται περίπου σε 20 εκατομμύρια εκτάρια έκταση που χρησιμοποιούμε διαφορετικά, όπου 10% μετατίθεται σε σχέση με άλλες χώρες ε, για ε, στόχους και χρήσεις παραγωγής. Ένας λόγος γι' αυτό ήταν ότι είχαμε συμφωνήσει κατά τη δεκαετία του 90 για την ανταγωνιστικότητα που είχε υποστεί πλήγματα όσον αφορά τα πρωτεϊνικά. Και γι' αυτό αυτός ήταν ο λόγος η φθηνή σόγια που πλημμύρισε τις αγορές μας. Είχαμε μείωση στα πρωτεϊνικά 30% όσον αφορά τα όσπρια και 3% μόνο της ευρωπαϊκής έκτασης ε, καλλιεργείται με πρωτεϊνούχα. Στη Γερμανία μάλιστα ένα μόνο της 100. Η ευρωπαϊκή παραγωγή έφτασε σε ένα κρίσιμο σημείο πλέον, όπου η έρευνα, η ανάπτυξη, ακριβώς όσον αφορά τα πρωτεϊνούχα στην Ευρώπη, τα πρωτεϊνούχα φυτά, διακυβεύονται αυτά. Εδώ πρέπει να ξεκινήσουμε ώστε να προαχθεί η παραγωγή των πρωτεϊνούχων, γιατί θα φτάσουμε σε ένα κατόφλι όπου θα υπονομεύεται πλέον και θα διακυβεύεται η παραγωγή μας και έτσι θα χάσουμε και τις θετικές επιπτώσεις που έχουν οι καλλιέργειες πρωτεϊνούχων στην γεωργία για όσον αφορά σκόπιμες επιπτώσεις. Υπάρχουν τεράστια δυναμικά για την ευρωπαϊκή παραγωγή και καλλιέργειες πρωτεϊνούχων. Ένα σημείο είχαμε αναφέρει. Ισότιμες ισοδίκες συνθήκες ανταγωνισμού πρέπει να διασφαλιστούν. Η συμφωνία Blair House πιστεύω εγώ, αμφισβητείται και πρέπει ίσω και να καταληθεί. Αυτό το οποίο όμω είναι σημαντικό για μα είναι τα πρωτεϊνούχα στο μέλλον, στη νέα διαμόρφωση τη ΚΑΠ, να διαδραματίσουν ένα σημαντικότερο, ένα κέριο ρόλο. Διότι πολλά θετικά σημεία σε σχέση με τη νέα ΚΑΠ συνενώνονται εδώ. Είναι σημαντικό λοιπόν και για την προστασία των υδάτινων πόρων και για την προστασία του περιβάλλοντος και για την βιοπικιλότητα. Και θέλω να αναφέρω ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα, οι καλλιέργειες αυτές ε, έχουν μεγάλη σημασία για την δέσμευση του διοξιδίου του άνθρακα και όσον αφορά και τα, το άζωτο θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ και γι' αυτό θα θέλαμε σε σχέση με αυτές τις καλλιέργειες αυτά, αυτές να αποτελέσουν ένα σταθερό στοιχείο της μελλοντική γεωργικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημαντικό όμω είναι για μας και αυτό έχει κέρια σημασία μείωση της εξάρτησής μας από τις εισαγωγές και διασφάλιση έτσι στο τέλος τέλος των ευρωπαϊκών παραγωγών χωρίς να υπάρχει εξάρτηση από εισαγω... των παραγωγών της Ευρώπης χωρίς να εξαρτώμαστε από εισαγωγές. Στην πρώτη θέση βρίσκεται σήμερα και εκείνα που σε σχέση με αυτό το θέμα έχουμε έναν ανταγωνιστή λοιπόν σε αυτόν τον τομέα. Αν όμως ε, τα θέσουμε αυτά στο σωστό επίπεδο πρέπει να δούμε κάποια σημεία πρέπει να φωτίσουμε τα οποία και να τα εξετάσουμε τα οποία έχουν ενταθεί στην έκθεση. Διευκολύνσεις για παράδειγμα εισαγωγών ε, προϊόντος σόγιας. Πρέπει εδώ να εισαχθεί μηδενική ανοχή. Πιστεύω ότι αυτό το στοιχείο μας δεν ανήκει σε αυτή την έκθεση. Και είναι μάλιστα και αντιπαραγωγικό αν ενταχθεί αυτό το, αυτό το στοιχείο ως παράγοντας στην δική μου έκθεση. Πρόκειται εδώ για την προαγωγή της ευρωπαϊκής παραγωγής πρωτεϊνούχων και όχι για την διευκόλυνση εισαγωγών από τρίτες χώρες. Να το αποσαφηνίσουμε αυτό σε σχέση με την έκθεση. Η έκθεση σε αυτό το σημείο πρέπει να ψηφιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να καταψηφιστούν αυτά τα στοιχεία, να μην ενταχθούν στην έκθεσή μου. Γιατί διαφορετικά θα είχα πρόβλημα να είναι η έκθεση στο όνομά μου και να εμπεριέχονται τέτοια στοιχεία. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε συνάδελφε Χόισλινγκ. Λοιπόν, ίσως μας εκπλήσει, αλλά και ευτυχώς παρότι έχει προχωρήσει ήδη η ώρα, δεν λέω της νύχτας αλλά του πρωινού, έχουμε δέκα συναδέλφους που έχουν εγγραφεί. Δεν είναι παραπάνω από αυτούς που είναι παρόντες. Πρώτη, θα λάβει τον λόγο η κυρία Μαγκίνες λοιπόν. Έχετε ένα λεπτό κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ Πρόεδρε, απλώς να πω στον εισηγητή μας ότι είναι πολύ καλή η έκθεση του και πολύ σωστά δίνει έμφαση στο ότι πρέπει να προσέξουμε τις εισαγωγές ε, τροφίμων για τις ποτενικές μας ανάγκες. Η σχέση μας εδώ με την Κίνα είναι σημαντική. Πρέπει τα θέματα να τα δούμε από την άποψη της επισητιστικής ασφάλειας. Γνωρίζω, Πρόεδρε, ότι εδώ μπορεί να μιλήσω περισσότερο από ό,τι θα θέλατε, διότι το ρολόι δεν έχει αρχίσει να μετράει σωστά. Τέλο πάντων, για του γενετικώ τροποποιημένου οργανισμού, όπω αναφέρονται στην έκθεση, ε, το εδώ και τώρα που απαιτεί αυτή η έκθεση, η άμεση ανάληψη ευθύνη και η μη έγκριση των γενετικώ τροποποιημένων οργανισμών είναι κάτι που απασχολεί του κτηνοτρόφου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να βρεθεί εδώ μια επιστημονική λύση και να προσέξουμε τι εξελίξει παγκοσμίω το θέμα αυτό. Αλλά και για τι πρωτενε είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα. Εφόσον εφαρμόζουμε του κανόνε που εδώ ισχύουν. Αλλά εφόσον κάποιε ζωικές πρωτεΐνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις ε, απαγορεύσαμε για σκοπού ανθρώπινη υγεία και ζωική ευζοία, πρέπει να σκεφτούμε πολύ προσεκτικά τι ποια θα είναι τα επόμενα βήματά μα. Γι' αυτό η έκθεση πολύ σωστά εντοπίζει ορισμένα από τα βασικά ζητήματα τη Ευρώπη για τα ερχόμενα χρόνια. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για τη γενεοδορία σας, κυρία. Στη συνέχεια θα λάβει τώρα τον λόγο ο κύριος Ταραμπέλα. Ένα λεπτό κύριε Ταραμπέλα. Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχήν και εγώ να ευχαριστήσω το διοικητή για την σημαντική του έκθεση παρά το γεγονός ότι έχω απογοητευτεί από την τελική του μορφή. Γι' αυτό και στην ε, αρμόδια επιτροπή είχα απόσχει από την ψηφοφορία, κατά την ψηφοφορία. Η έκθεση τελικά παραμορφώθηκε από τις ε, τροπολογίες για, με τρόπο που δεν λύνει το πρόβλημα έλλειψης πρωτεϊνών στην Ένωση. Αλλά μην ξαναρχίσουμε εδώ αυτή τη συζήτηση. Η καλλιέργεια πρωτεϊνούχων στην Ευρώπη για τη μείωση της εξάρτησής μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό θέμα γιατί πρέπει να μας ανησυχήσει όλους. Και εγώ συμφωνώ με αυτά που υπόθηκαν για τη συμφωνία του Δερχάους. Οι συμφωνίες αυτές είναι σε πλήρη αντίθεση με το πρωτόκολλο του Κιώτου για την κλιματική θέρμανση. Εξάλλου, οι, τα πρωτεϊνούχα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται γενικότερα στο γενικότερο κύκλο των καλλιεργειών. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Φερέιρα παρακαλώ θα λάβει τον λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το έλλειμμα πρωτεϊνούχων φυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία εκδήλωση ακόμα των ανισοτήτων της εντατικής παραγωγής της ΚΑΠΑ αυτή η τάση έχει άμεσες επιπτώσεις στον τομέα της ασφάλειας, της επιστημιστική ασφάλειας και της ποιότητας της επιστημιστική ασφάλειας των πολιτών. Έχει ιδιαίτερα πλήττει τους ε, παραγωγούς ε, που ασχολούνται με την κτηνοτροφία. Ένα σύνολο μέτρων πρέπει να ληφθούν υπόψη υπέρ των πρωτενούχων, υπέρ τη τοπική παραγωγή. και σε σύντομες αλυσίδες παραγωγής ώστε να μειωθούν σταδιακά οι εισαγωγές. Αυτά τα μέτρα μπορούν να συμπεριλαμβάνουν εξειδικευμένα μέτρα σε σχέση με την ανακύκλωση παραγωγών, έρευνα και ανάπτυξη και άλλα συναφή μέτρα. Αυτό το πρόβλημα δεν μπορεί να είναι πρόσχημα για τη δημιουργία άλλων μεγαλύτερων προβλημάτων. Έτσι δεν μπορεί να ισχύσει οποιαδήποτε ε, παρέμβαση όσον αφορά την μηδενική ανοχή ή την πρόληψη, την αρχή της εφαρμογής τη πρόληψης εξαντλήσατε τον χρόνο. Δεν σε ακολουθούσαν ε, οι, εισαγωγοί, οι διερμηνείς σε αυτό το ε, δρόμο ταχύτητας ε, στην τελική ευθεία. Η κυρία Ντότς παρακαλώ. Uh, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή για αυτή τη σημαντική έκθεση. Εδώ η τιμές των τροφίμων και απαγορεύσεις κάποιων καλλιεργειών δείχνουν πόσο εκτεθειμένη μπορεί να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προμήθεια ορισμένων πρώτων υλών για το κτηνοτροφικό τομέα. Ζωτική σημασία αυτά ε, και οι εκλογέ μου στη δική μου την εκλογική περιφέρεια, ιδίω στον τομέα των εκτροφή χείρων, βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση. Εδώ λοιπόν ο εισηγητή νομίζω σωστά εντοπίζει ότι η Ευρώπη πρέπει, οφείλει να κινηθεί προ μία λύση σε σχέση με τη μηδενική ανοχή. Την περασμένη μόλι εβδομάδα μιλούσα σε εκλογή μου στην εκλογική μου περιφέρεια, οι οποίοι είναι εισαγωγή ζωοτροφών και έλεγαν ότι για την ώρα μόνο σε πολιτικά εμπόδια φαίνεται να προσκρούν με τους νέους κανόνες. Δεν είναι πραγματικές οι λύσεις που προσφέρονται. Πραγματικές λύσεις μας ζητάνε σε σχέση με τη μηδενική ανοχή. Στη συνέχεια κύριε Νταντάν παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ ως κοιόδης εισηγητής της ομάδας μου να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη συνεργασία που είχαμε. Το θέμα αυτό αγαπητοί συνάδελφοι έχει στρατηγική σημασία. Έναν αριθμό θα σας δώσω. Μιλήσαμε για την Κίνα. Το 2010 οι Κινέζοι αγόρασαν 49% των ζωοτροφών σόγιας και οι προβλέψεις για το 2011 είναι να αγοράσουν το 55% της παγκόσμιας αγοράς. Επομένως τίθεται εδώ ένα θέμα εξάρτησης της Ένωσης. Μπορεί κανείς να φανταστεί ποτέ ότι η περιοχή εκείνη με τόσο εντατική γεωργία μπορεί κάποτε να πάψει να αγοράζει σόγια. Η χώρα μου δημιούργησε μια πολιτική σύμφωνα με το άρθρο 68 που απέδειξε ότι είναι ευέλικτη η γεωργία μας και... Ο κύριος Ταμπασδής συνέχεια παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Όσο αρμόδιος ε, για τη σοσιαλιστική ομάδα και ως συντάκτης νομοδότησης, ε, της νομοδότησης για την Επιτροπή Περιβάλλοντος δράτω με τις να συγχαρώ τον κύριο Χόισλινγκ τον ευχαριστώ για μια εξαιρετική συνεργασία που είχαμε. Είναι καλή αυτή η έκθεση. Κάνουμε τον λόγο για το γεγονό ότι έχουμε έλλειμμα πρωτεϊνούχων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πραγματικό κίνδυνο για την κτηνοτροφία και την ε, διατροφή των ε, ζώων στην κτηνοτροφία στην Ευρώπη. Οι κλιματικέ ε, συνθήκε. Τι γίνεται και με το σύστημα τη υποστήριξη. Δεν δίνουμε επαρκή υποστήριξη σε σχέση με τα πρωτεϊνούχα δυστυχώ. Μία πτυχή που είναι σημαντική θα ήθελα να επιστήσω στην προσοχή σα Μόνο κυρία, κυρία Δαμανάκη, ως Επιτρόπου, είναι ανάγκη άμεσα να δράσετε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να αντιμετωπίσετε τα θέματα ε, ζωικών ε, πρωτεϊνών και κάνουμε λόγο εδώ για τα πουλερικά και τα, και τα Υπάρχει ανάγκη να εξεταστεί αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σικέρσκης στη συνέχεια παρακαλώ. Σας ευχαριστώ η κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδήγησε σε αυτή την κατάσταση όπου βλέπουμε ότι τα πρωτενούχα και η παραγωγή τους δεν είναι πλέον κερδοφόρα και το έλλειμμα πρωτενούχων δείχνει ότι θα έπρεπε να προβληματιστούμε σε βάθος για τις πολιτικές μας. Αυτή τη στιγμή στην ευρωπαϊκή αγορά έχουμε σόγια που εισάγεται αποκλειστικά από την Βραζιλία, την Αργεντινή, τη ΣΥΠΑ κτλ. Και βλέπουμε ότι πρόκειται για σόγια για φυτά που έχουν, ε, είναι γενετικά τροποποιημένα και ε, έχουν προσιτές φθηνές τιμές. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η διαθεσιμότητα και η προσπελασιμότητα των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών για τις ευρωπαϊκές αγορές. Δεν είμαστε όμως συνεπείς. Αφενός από τη μία πλευρά κάνουμε λόγο για απαγόρευση ε, γενετικά τροποποιημένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη πλευρά έχουμε γενετικά τροποποιημένη σόγια που εισάγεται από τρίτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι γίνεται εδώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα ολοκληρώσουμε τη συζήτηση με την παρέμβαση της κυρίας Βέσλον. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστούμε και τον εισηγητή ε, για την ε, πολύ καλά ε, συνταγμένη εκθεσή του. Είναι πραγματικά ξεχωρίζει σχέση με άλλε εκθέσει που έχουμε συζητήσει εδώ στην Ολομέλεια. Μιλώντα για του κινητικό τροποποιημένου λοιπόν οργανισμού και την σχετική απαγόρευση, να πω ότι στην έκθεση αυτή δεν τονίζεται αρκετά το θέμα αυτό, δεν βρίσκεται στη σωστή του θέση. Επίσης δεν αναφέρονται κάποιες, κάποια κλιματικά στοιχεία θετικά με το σωστό τρόπο. Δηλαδή ε, κάποιες καλλιέργειες πρωτεϊνών στην Ευρώπη υπάρχουν και χρειάζονται. Όμως το θέμα είναι να δούμε τις ανάγκες κατανάλωσης που αυξάνονται. Και επίσης, να μην ξεχνάμε τόσο περισσότερο κρέα καταναλώνουμε, τόσο περισσότερο κάνουμε κακό στο κλίμα και στις καλλιέργειες, ε, τι κλασικέ. Αυτό λοιπόν πρέπει να επιλύσουμε κυρίω. Ποιο είναι το μέλος αυτών των. Σα ευχαριστούμε, κυρία Βέσλοντ. Είχαμε ξεχάσει και ζητώ συγγνώμη τον κύριο Σον Κέλλη, με τον οποίο θα ολοκληρώσουμε αυτό τον γύρο παρεμβάσεων. Ο κύριο Κέλλη. Ε, ε, Ευχαριστώ. Όπως σωστά αναφέρει ο κύριος ε, Χόσλινγκ Πολλές φορές εδώ έχουμε να κάνουμε με καταστάσεις ε, που μας σκανδαλίζουν, διότι η παραγωγή πρωτεϊνών στην Ευρώπη είναι τόσο ανεπαρκής που μας δείχνει ότι είμαστε εξαρτημένοι από εισαγόμενα προϊόντα. Αυτό προφανώς είναι αλληλένδετο και με την παραγωγή γεωργικών ε, προϊόντων και με τα κοπάδια των ζώων. Την κτηνοτροφία λοιπόν. Εδώ ένα θέμα <clears throat> είναι η αυτονομία μας σε σχέση με τις εισαγωγέ. Αυτό είναι πολύ εύκολο να το λέμε, αλλά πρέπει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην πράξη. Επίσης, τον το, ε, μεταξύ των στόχων της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ, πρέπει να σκεφτούμε τι θα κάνουμε για να είμαστε ε, ε, αυτάρκεις. Ευχαριστούμε κύριε Κέλλη. Μια και ολοκληρώθηκε εδώ ο γύρο των παρεμβάσεων των συναδέλφων που παρενέβησαν, θα δώσουμε τον λόγο στην Επίτροπο, την κυρία Δαμανάκη, για να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Κυρία Δαμανάκη, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μία βιώσιμη προμήθεια πρωτεϊνών είναι ουσιώδης για τον κτηνοτροφικό μας τομέα. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας που έθεσαν το σημαντικό αυτό θέμα ενώπιον μας. Η έκθεσή σας γίνεται ευπρόσδεκτη από μας για τα πλαίσια της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ προς το 2020. Όπως ξέρετε η Κομισιόν προτίθεται να κάνει προτάσεις σχετικά το φθινόπωρο. Θα ήθελα να τονίσω ότι η εσωτερική παραγωγή πρωτεϊνών έχει αυξηθεί με τα υποπροϊόντα των βιοκαυσίμων. Οι εθανόλοι ιδιαίτερα αντιπροσωπεύουν τώρα όλα αυτά το 22% της κατανάλωσης πρωτεϊνών στην Ένωση σε σύγκριση με 12 μόνο της 100 πριν από 5 χρόνια. Η στήριξη των γεωργών είναι από τις κυριότερες ιδέες της εκθεσής σας όπως ξέρετε και εμείς συζητάμε την εκθέση αυτή για το πρασίνισμα της παραγωγής δεχόμαστε λοιπόν την ιδέα σας για τη βιώσιμη παραγωγή γιατί βλέπω και εδώ πρόσθετες ευκαιρίες για να υπάρξει περισσότερη συνέργεια για καλύτερη διαχείριση όμως οποιοδήποτε πρασίνισμα των πληρωμών δεν θα έπρεπε να αφισβητήσει την αποσύνδεση από τις επιχορηγήσεις. Η ιδέα αυτή είναι βασική για την ε, κατεύθυνση που έχουμε δώσει στις προηγούμενες μεταρρυθμίσεις. Θα ήθελα να τονίσω ότι πολλές χώρες μέλη αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούν τη δυνατότητα σύνδεσης άμεσων επιχορηγήσεων με περιβαλλοντολογικούς στόχους για την παραγωγή πρωτεϊνούχων. Επίσης τονίζω ότι η αύξηση της παραγωγής σόγιας στην Ένωση θα σημάνει μάλλον μείωση της, ανάλογη μείωση της παραγωγής δημητριακών, γιατί δεν έχουμε περιόριστες γέες. Τέλος θα ήθελα να τονίσω άλλους δύο τομείς όπου η πολιτική της Ένωσης μπορεί να συμβάλλει. Η έρευνα και η περιφερειακή ανάπτυξη μπορούν και τα δύο αυτά να αποτελέσουν μια καλή ευκαιρία διαφοροποίηση των πηγών πρωτεϊνούχων μας. Παραδείγματο χάρην καλύτερη χρήση της σοδιάς και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 Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Επίτροπε. Και ολοκληρώνεται έτσι η συζήτηση. Και αύριο το μεσημέρι 12.00 θα ψηφίσουμε την αντίστοιχη πρόταση ψηφίσματος. Συνάδελφοι, η επόμενη συνεδρία θα γίνει αύριο, θα διεξαχθεί αύριο 3η 8 Μαρτίου από τις 9